Παρακαλώ καθίστε. Τα χτεσινά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι διαθέσιμα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Θα, θα εγκριθούν. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και τις Επιτροπή για τα διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία. Το λόγο έχει για το Συμβούλιο η κυρία Γκέρι. Bien, señorías, Κυρίες και κύριοι, δια... είδαμε αυτό το ωραίο θέαμα, όμορφο θέαμα. Θα σας παρακαλούσα, αν γίνεται για την καλή τη λειτουργία της ε, Συνόδου, να καθίσετε και να μην χρησιμοποιείτε πλέον οπτικά σήματα ξένα σε σχέση με την Ολομέλεια. Κύριε Γεώργη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, επιτρέψτε μου καταρχά να πω ότι χαίρο που μπορούμε να συνεχίσουμε εδώ τις συζητήσεις που είχαμε ξεκινήσει τον περασμένο μήνα που δείχνει πόσο σοβαρό είναι το θέμα αλλά και πέραν των συναισθηματικών αντιδράσεων που όλοι ε, είχαμε λόγω των, των γεγονότων στην Ιαπωνία χρειάζεται να υπάρξει μια συνολική αντίδραση. Επιτρέψτε μου καταρχά να επιβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να βοηθήσουμε συγκεκριμένα και μόνιμα τον Ιαπωνικό λαό είτε σε υπομορφή ανθρωπιστική είτε υπομορφή παροχής βοήθειας ε, πυρηνικών ειδικών. Το Συμβούλιο στις 25 Μαρτίου το υπογράμμισε. Να επιστήσω επίσης την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Ουγγρική Προεδρία ε, αμελητή αντέδρασε στις εξελίξεις μετά την καταστροφή στην Ιαπωνία, ιδίως το κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος. Επίσης, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχουν συζητήσεις για θέματα πυρηνική, πυρηνικού κινδύνου που θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν. Στην Ευρώπη πάνω από 25 χρόνια ισχύει ένα νομοθετικό πλαίσιο δεσμευτικά, δεσμευτικό νομικά που επικαιροποιούμε συνεχώς. Θέλω να αναφερθώ ιδίω εδώ στην οδηγία του 2009 για την πυρηνική ασφάλεια. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό διότι η πυρηνική ασφάλεια είναι μια μόνιμη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας προσπαθούμε να αντλήσουμε τα διδάγματα ιδίως ε, μετά από γεγονότα όπως αυτά που είδαμε για τη Φουκουσίμα και να παρακολουθούμε και να επαληθεύουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επιπλέον ότι οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό μορφή απάντησης στο στο συμβάν έχει ως στόχο την τελειοποίηση και την εξασφάλιση του νομοθετικού πλαισίου. Οι αντιδράσεις της Ένωσης στηρίζονται στην ιδέα ότι ο κίνδυνος που περιβάλλει τους πυρηνικούς σταθμούς θα πρέπει να αντιμετωπίζει ε, ελέγχους αντίστασης, δηλαδή τα stress test. Επιπλέον, τα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι γνώσεις των ειδικών στον τομέα αυτό θα πρέπει να επιτρέπουν την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος. Η ομάδα και τα μέλη της ομάδας υπεύθυνη για την ε, νομοθεσία σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να επεξεργαστεί μέχρι τα μέσα Μαΐου ένα, μια σειρά στοιχείων που θα μας επιτρέπουν θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση αυτή. Πολλά κράτη-μέλη, πολλά κράτη ειδικότερα που χρησιμοποιούν πυρηνικούς σταθμούς, ήδη έλαβαν τις πρώτες αποφάσεις για τον έλεγχο ασφάλειας των σταθμών αυτών. Μέχρι το τέλος του έτους προφανώς θα μπορέσουμε να ε, αντλήσουμε τα πρώτα διδάγματα. Επιπλέον κάτι που, επί του οποίου συμφωνεί και η κοινή γνώμη και η Επιτροπή είναι ακριβώς αυτό. Βάσει των τελευταίων δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο νομοθετικού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παληθεύσει και να ελέγξει όλες τις ρυθμίσεις που συνοδεύουν την υλοποίηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ώστε να το να ολοκληρωθεί όσο περισσότερο γίνεται και να τελειοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό της ε, του, κανονιστικού πλαισίου συνεχίζονται κάποιες εξελίξεις, ε, κάποιες ε, προτάσεις, ενώ εξετάζουμε και την πρόταση οδηγία για την επεξεργασία των ε, ραδιενεργών ε, καταλήπων, ιδίως την εξέλιξη των, των, ε, των αποβλήτων αυτών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τρίτον, μια έκκληση προς τις τρίτες χώρες γείτονες της Ένωσης να μετάσχουν και αυτές στο ίδιο εγχείρημα, δείχνοντα υπευθυνότητα και μέρημνα για την ασφάλεια. Αυτά δεν περιορίζονται βέβαια μόνο στην πυρηνική ενέργεια. Ανεξάρτητα από το ποσοστό ενέργειας που παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει ε, εφοδιασμός της Ένωσης σωστός και να μην υπάρξει κίνδυνος ε, για την ασφάλεια των ατόμων. Επίσης, θα πρέπει την ασφάλεια στην Ευρώπη να τη δούμε και από την οπτική γωνία της χρήσης από πλευράς κατών μελών ε, του ενεργειακού μίξ που είναι ένα δικαίωμα των κρατών μελών. Αυτό το έχουμε δηλώσει. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ταυτόχρονα μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματα που έχουμε κοινά, την πολιτική ενέργειας. Φέτος θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε την ε, το μέλλον της ενέργειας εν ώψη του 2050 και να δούμε πώς θα συνοδεύουμε τα μέτρα για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και να επιτύχουμε όλους τους άλλους στόχους ανταγωνιστικότητας ιδίως. Πέραν της ε, ελευθερίας επιλογής του ενεργειακού μίξ των κρατών μελών και τους στόχους της ενιαίας αγοράς, πρέπει να λάβουμε υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών ε, από, ε, από... από την ενεργειακή πολιτική και τις συναφείς αποφάσεις. Θα πρέπει ιδίω να υιοθετήσουμε τις συνέπειες ε, στις επενδύσεις στην ενέργεια και άρα να δούμε ότι παράλληλα με την παραγωγή ενέργειας που εξαρτάται κατά 30% από την πυρηνική ενέργεια, κανένα από τα 14 κράτη-μέλη που έχουν πυρηνικούς σταθμούς δεν θα μπορούν να κλείσουν τους σταθμούς αυτούς χωρίς να ζητήσουν την άποψη των υπόλοιπων κρατών μελών για να εξετάσουν τις εναλλακτικέ λύσεις, ιδίως ό,τι αφορά τα δίκτυα και την εξάρτηση. Από την οπτική αυτή γωνία, οι Υπουργοί Ενέργειας στην άτυπη συνάντησή τους τον Μάιο θα ασχοληθούν με το ζήτημα, θα προβούν δηλαδή σε μια ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες να προχωρήσουμε από κοινού. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό επίσης, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιλογές για να εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων επιλογών. Είμαι πεπισμένη ότι οι συζητήσεις που έχουμε εδώ σήμερα θα συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Το λόγο έχει τώρα, ευχαριστώ την Υπουργό, το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Έτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ο φρικτός σεισμός της 11ης Μαρτίου, το τσουνάμι που επέφερε και μετά το πυρηνικό ατύχημα με σημαντικές βλάβες στα διάφορα μπλοκ, στους διάφορους αντιδραστήρες που ακόμη μέχρι τώρα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς ούτε φαίνεται να υπάρχει ούτε ε, ε, διαφαίνεται το τέλος των προσπαθειών όλα αυτά μας απασχολούν σε σχέση με την ασφάλεια την ενέργεια και την διαχείριση της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Ήδη λοιπόν στις 11 Μαρτίου προσκαλέσαμε και στις 15 Μαρτίου διεξαγάγαμε συνεδρίαση ομάδας υψηλού επίπεδου με εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των κατασκευαστών πυρηνικών σταθμών αλλά και εκπροσώπων της ε, οικονομίας της ενέργειας και συζητήσαμε σε προπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που κατόπιν μετά από λίγες ημέρες έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει δοκιμασία αντοχής με αυστηρότατα κριτήρια. Από τότε επεξεργαζόμαστε τα κριτήρια της δοκιμασίας αυτής. Η Γενική Διεύθυνση, εγώ προσωπικά μαζί με τις αρχές εποπτείας, συντάσσουμε τις ημέρες αυτές κατάλογο κριτηρίων δοκιμασίας που πριν λάβει την τελική του μορφή θα υποβληθεί και σε εσάς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα είναι διαφανής και για την κοινή γνώμη. Αφενός λοιπόν πρόκειται για τις επιπτώσεις λόγω κινδύνων σεισμών ή πλημμυρών, κυρίως στον Ατλαντικό, για τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη, για τις επιπτώσεις στο ίδιο το εργοστάσιο, δηλαδή πώς μπορεί να παραμείνει ασφαλής η λειτουργία των συστημάτων ψήξεως, επίσης τα συστήματα παραγωγής ενέργειας για το ίδιο το εργοστάσιο σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του, επίσης για ενδεχόμενα ατυχημάτων ή άλλων παραγόντων όπως πτώσεως αεροσκαφών κλπ. Όλα αυτά λοιπόν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούμε ότι μετά, μέσα Μαΐου μάλλον στα πλαίσια της Διεθνούς Αρχής Εποπτείας των Πυρηνικών Εργοστασιών θα μπορέσει να δοθεί τελική μορφή στο έγγραφο και στα μέσα του έτους και μέχρι τα τέλη του έτους θα μπορέσουν να διεξαχθούν πλήρεις δοκιμασίες με τον στόχο να είναι εγγυημένα τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας των ευρωπαϊκών πυρηνικών αντιδραστήρων. Ε, λάβαμε επαφή με τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Κοινοπολιτείας, της Ουκρανίας. Αυτές τις επαφές θα τις συνεχίσουμε, θα τις επεκτείνουμε και στην Ελβετία και επίσης με την Αρμενία, αλλά και με χώρες οι οποίες σχεδιάζουν την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων όπως η Τουρκία και η Λευκορωσία. Όλα αυτά με τον στόχο αυτά τα υψηλότατα επίπεδα ασφαλείας, τα κριτήρια να διασφαλίζονται και στις χώρες άμεσης γειτονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα για το λεγόμενο μείγμα ενέργειας και επομένως και για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και άρα και για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες ή άλλες τεχνολογίες ε, είναι ανήκει στις χώρες μέλη. Τις τελευταίες ημέρες φάνηκε ότι οι χώρες μέλη έχουν ενδιαφέρον να διατηρήσουν την αρμοδιότητα αυτή. Άρα, εν τέλει, η απόφαση για την χρήση της πυρηνικής ενέργειας στα πλαίσια των συνθήκων δεν μπορεί να εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι δοκιμασίες ασφάλειας στις οποίες θα συμμετάσχουν όλοι μου φαίνεται ότι πρέπει και μπορεί να είναι ο κοινό παρονομαστή όλων των χωρών μελών, είτε διαθέτουν πυρηνικά εργοστάσια, είτε τα απορρίπτουν. Η Γαλλία λαμβάνει το ρεύμα της κατά 76% από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η Αυστρία 0%. Άλλες χώρες σε ποικίλα ποσοστά. Η Γερμανία εξετάζει την μείωση της διάρκειας ε, λειτουργίας των ε, πυρηνικών αντιδραστήρων. Η Ιταλία και η Πολωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο η Ιταλία να ξαναμπεί στην πυρηνική ενέργεια, η Πολωνία για πρώτη φορά. Εκτός από τα τσέκ αυτά, βασιζόμαστε και στην εφαρμογή, στην μεταφορά μάλλον της ε, σχετικής οδηγίας στα εθνικά δίκαια μέχρι τον Ιούλιο φέτος. Μέχρι τώρα είχαμε σκοπό το 2014 να κάνουμε αξιολόγηση των ε, ε, διατάξεων ασφαλείας, αλλά θα προτάξουμε την προσπάθεια αυτή. Μέχρι το τέλος του 2012 θα σας υποβάλουμε έγγραφα σχετικά με αρχές που πρέπει να δημιουργηθούν με την εφαρμογή των κριτηρίων των αρχών ασφαλείας κλπ. Υπάρχουν και τα σχετικά εγγραφά για τα πυρηνικά κατάλοιπα τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητούνται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και αυτά αποτελούν συμβολή στα περαιτέρω βήματα και μέτρα για την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών επιπέδων ασφαλείας. Γνωρίζουμε ότι μετά από τη δοκιμασία αντοχής θα προχωρήσουν εθελοντικώ σε λήψη μέτρων οι χώρε μέλη. Δεν θα είναι αναγκαστικά, αναγκαστικέ οι προτάσει αυτέ. Τα απαραίτητα μέτρα θα προταθούν από του εμπειρογνώμονε, θα γίνουν δεκτά από τι χώρε μέλη και θα εφαρμοστούν στου ενδεχόμενου πυρηνικού του αντιδραστήρε. Θα σας ενημερώσουμε ξανά περί τα μέσα Μαΐου σχετικά με το σχέδιο για τις δοκιμασίες αντοχής και για τις σχετικές προφορίες που θα έχουμε λάβει από τις εργασίες της ομάδας εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στους αγωγητές των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Βότμαν Κόλ. Καλημέρα σας Πρόεδρε, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Έτσιγκερ, ο οποίος αμέσως αντέδρασε στο θέμα αυτό της πυρηνικής ενέργειας αμέσως μετά την ε, μεγάλη καταστροφή στην Ιαπωνία, που το κρίνουμε πολύ σημαντικό για την ασφάλεια όλων των πολιτών μας. Ε, η πυρηνική αυτή καταστροφή στην ε, Ιαπωνία δείχνει ότι πρέπει να αλλάξουμε στάσεις στο θέμα τη πυρηνική ασφάλεια. Τουλάχιστον να αναθεωρήσουμε τι θέσει μα. Και εδώ έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξαρτώμεθα ημέν από του δε στα θέματα τη πυρηνική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ελέγχους δοκιμές πυρηνικής αντοχής στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, ασφάλειας δηλαδή, σε, όλους τους, σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης και απαιτείται να δίδονται στο κοινό οι σχετικές εκθέσεις, να δημοσιοποιούνται. Ελπίζω κύριο Έτιγκερ να ακολουθήσετε μία προσέγγιση σε εναρμονισμένη συνεργασία με τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλιστεί η βάση που χρειάζεται και αν τυχόν κάποια πυρηνική εγκατάσταση αποδειχθεί ότι δεν περνάει την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για το τεστ αντοχής, τότε θα πρέπει να αναλαμβάνονται αμέσως από το αρμόδιο κράτος μέλος τα μέτρα που απαιτούνται για προσωρινή ή και μόνιμη πάυση λειτουργίας και Πιστεύω αυτό πρέπει να ισχύσει, να το διεκδικήσουμε και για τις πυρηνικέ εγκαταστάσεις που έχουμε στα σύνορα της Ευρώπης, από την άλλη πλευρά των σύνορων δηλαδή, και που είναι ακόμη πιο επικίνδυνες πολλές φορές για την ασφαλεία μας. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είμαστε θέση να αξιολογούμε τους κινδύνους ε, μέσα στου σωστού όρου. Η πυρηνική ενέργεια είναι μια πηγή την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, δεν μπορούμε ανεφετέρου δηλαδή να την πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Μα εξασφαλίζει σημαντική ποσότητα ηλεκτρική ενέργεια, μα βοηθάει να μειώσουμε τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Παράλληλα όμω θα πρέπει να ανοίξουμε και τα μάτια προ το μέλλον και άρα πρέπει να στραφούμε και προ ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και να κάνουμε την προσπάθεια που χρειάζεται για να τι ενισχύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βόρτμαν Κόλ. Τώρα για δύο λεπτά η κυρία Ουλίσκοκ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η πυρηνική είναι μια πηγή ενέργειας που διαφοροποιείται από τις λοιπές. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορεί να επιφέρει τεράστιες ζημιές στη χώρα, το έδαφος δηλαδή, αλλά και τους πολίτες της ε, και μάλιστα για πολλές γενναίες. Στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας τα θέματα της ασφάλειας νομίζω ότι χάνουν συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι θα, μεταφραστούν σε, θα μετατραπούν σε κοινέ και συνενετικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, δεν γνωρίζει σύνορα εθνικά, όπως δεν γνωρίζει σύνορα ευρωπαϊκά η πυρηνική ενέργεια. Και γι' αυτό ο διάλογος για την πυρηνική ενέργεια και την πυρηνική ασφάλεια έχει ευρύτατη εμβέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται στο δυνατόν πιο εναρμονισμένε και πιο ομοιόμορφε ή κοινέ αποφάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις θέσεις μας ως προς την ίδια τη χρήση των πυρηνικών, έχοντας πάντοτε υπόψη μέσο και μάκρο πρόθεσμα και ως κύριο γνώμονα την ασφάλεια. Υπάρχει ασφαλώ το επιχείρημα ότι δεν έχουμε το ενεργειακό εκείνο μείγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να, με, να εγκαταλείψουμε ε, ταχύτατα την πυρηνική ενέργεια και να στραφούμε προς άλλες ε, πηγές. Όμως πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερο και να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σημείο καμπής, έχουμε να κάνουμε με, μια, με ένα ιστορικό σημείο το οποίο θα μας υποχρεώσει να μεταστρέψουμε το βλέμμα προς τη βιωσιμότητα, προς μια στρατηγική που θα μας επιτρέψει σε βράχη, μέσο ή και μακροπρόθεσμο ορίζοντα να κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια. Ευχαριστούμε κυρία Ουλσκοκ για του φιλελεύθερου και δημοκράτες. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Εκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι εξελίξη στην Ιαπωνία δεν έδειξε μόνο το πρόβλημα στους αντιδραστήρες της, της Ιαπωνίας αλλά και τα προβλήματα ευρύτερα των πυρηνικών σταθμών. Πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν σήμερα για την πυρηνική ασφαλεία στην Ευρώπη. Είναι αναγκαίο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να επανεξετάσει την προσέγγιση της προς την πυρηνική ασφάλεια. Οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες θεωρούν ότι οι προτάσει του Συμβουλίου παρά είναι Δεν θα έπρεπε να ε, ελέγξουμε τεχνολογία και τοποθέτηση, αλλά όλη την κουλτούρα ασφάλειας και την, την, την ετοιμότητά μας να ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστροφές πολύ, πολύ, πολύ μορφές είναι εξίσου ζωτικό να γίνουν υποχρεωτικοί έλεγχοι και με συγκεκριμένα κοινά αυστηρά κοινοτικά κριτήρια. Είναι προφανές σε όλου ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε στις ε, κυβερνήσει και τι εθνικέ αρχές την εποπτεία τους. Ε, τα stress test θα έπρεπε να διεξάγονται από ανεξάρτητους ειδικού με πλήρη διαφάνεια πρέπει να δημοσιεύονται όλα τα δεδομένα κατόπιν πρωτοβουλία τη Επιτροπή. Σήμερα αυτή είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση στην τεχνολογία αυτή. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρη, ολοκληρωμένη αναθεώρηση τη ε, νομοθεσία για την ποινική ασφάλεια, ε, με τον ε, δεχόμενη, δεχόμενη ευρωπαϊκά στάνταρ και απαιτήσει. αυτό είναι η ευθύνη τη Επιτροπή, αλλά και του Συμβουλίου να προωθήσει και να αναλάβει τι ευθύνε. Εν τέλει, είναι ουσιώδε να μάθουμε τα διδάγματα και για εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια και για την ενεργειακή απόδοση. Και καιρό είναι να αποφασίσουμε για δεσμευτικού στόχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους και Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία και για δυόμιση λεπτά η κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ. Κύριε Πέτινια, γνωρίζετε ότι δυσπιστώ απέναντι στα τεστ αντοχής. Και θα σας πω γιατί. Θεωρώ ότι ο ορισμός των κριτηρίων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων δεν μπορούν να παραμείνουν στα χέρια των εθνικών αρχών και των αρχών εποπτείας που ήταν αρμόδιες μέχρι τώρα μόνο για την εποπτεία και την εξέταση των πυρηνικών εργοστασίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι οποίοι θα δώσουν οι μεν στους δε πιστοποιητικά ασφαλείας για τα δίθεν ασφαλή πυρηνικά τους εργοστάσια. Ή θεωρείται σοβαρά ότι οι εθνικές αρχές εποπτείας θα καταλήξουν ξαφνικά στο συμπέρασμα ότι μέχρι τώρα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και είχαν φανεί υπερβολικά ανεκτικές. Δεν το πιστεύω αυτό κύριε Φέτιγκερ και ούτε μου έχετε εξηγήσει πώς θα επιτύχετε να υπάρξει πλήρης ανεξαρτησία τώρα ο δε εθελοντικός χαρακτήρας των δοκιμασιών αντοχής είναι άλλη μια απόδειξη για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά αυτά τα τεστ όσο θα θέλατε εσείς. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν σωστά με την πρόσβαση σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, με την διασφάλιση ότι θα ελεγχθούν τα πάντα και όχι ότι θα γίνουν μοναχά μελέτες επί χάρτου αυτό που εννοούσα προηγουμένως όταν δηλαδή οι ίδιοι θα δίνουν στους γνωστούς τους γιατί είναι γνωστοί μεταξύ τους όλοι οι υπεύθυνοι. Εμείς οι πράσινοι αναμένουμε η δοκιμασία, οι δοκιμασίες αντοχής να γίνουν με τέτοιον τρόπο ώστε να φανεί καθαρά ποια εργοστάσια δεν μπορούν να γίνουν πλέον ανοιχτά, ανεκτά, συγγνώμη, ποια πρέπει να καταλήψουν το δίκτυο ευθύ αμέσω οι δοκιμασίες αντοχής θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση για ένα χρονοδιάγραμμα κλεισίματος που ας αρχίσει τώρα και ας φτάσει μέχρι το 2025 αν θέλετε όπου στην Ευρώπη θα πρέπει να κλείσει και το τελευταίο εργοστάσιο. Θα σας παρακαλέσω για ένα πράγμα κύριε Έτιγκερ. Τελευταία δώσατε πολλές συνεντεύξεις, δηλώσατε για παράδειγμα στην Γερμανία ότι γνωρίζετε ήδη τώρα ποια πυρηνικά εργοστάσια δεν πρόκειται να περάσουν τι δοκιμασίε αντοχής. Ή είπατε τέλο πάντων ότι ορισμένα από αυτά δεν πρόκειται. Μα πέστε τα, πέστε τα με το όνομά του αν πρόκειται για το Φέσενχάιμ. Ένα εργοστάσιο το οποίο δεν είναι εξασφαλισμένο ούτε απέναντι σε πλημμύρε από τον ποταμό Ρήνο, ούτε απέναντι σε ενδεχόμενα σεισμών. Πέστε λοιπόν ποια είναι τα επικίνδυνα εργοστάσια. Μόνο αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε κάποια εμπιστοσύνη στην πολιτική σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Χάρμς για τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και για 1,5 λεπτό κύριο Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστώ την Προεδρεύουσα και τον Επιτροπό για τις ε, δηλώσεις τους. Το μέτρο που ακολούθησαν στη διατύπωση είναι σε ευθύ αντίθεση με αυτά που ακούμε από άλλους εδώ μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μετά τις ε, εξελίξεις στην Ιαπωνία και το νέο σχεδιασμό που βλέπουμε στην Ευρώπη που έχουμε στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όπω υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο μέγεθο του κινδύνου που αντιμετωπίζει καθημερινά η Ιαπωνία και η Δυτική Ευρώπη από την άλλη πλευρά. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε, ε, βέβαιοι ασφαλώ για το τι έχει πραγματικά συμβεί πριν αναλάβουμε κάποια μέτρα ενδεχομένω για την αναθεώρηση του τι πράττουμε και τι σκοπεύουμε να πράξουμε. Οι σύγχρονοι αντιδραστήρε που σχεδιάζονται τώρα έχουν ε, τη δυνατότητα να αντισταθούν σε μεγάλου κινδύνου που ήταν μάλιστα αδιανόητοι πριν από 20-30 χρόνια. Και βλέπω κυρία Χάρμς ότι συμφωνείτε μαζί μου. Κυρία Χάρμς χωρίς μικρόφωνο. Υπήρξατε αγενείς εκτός μικροφώνου. Κυρία Χάρμς μου αφαιρείτε από το χρόνο ομιλίας μου. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση για δικαιοστάσιο και το προτείνω διότι θα σήμαινε αυτό μια υπερβολική σπουδή χωρί να γνωρίζουμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Όχι, πρέπει να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί πριν να αναλάβουμε κάποιο μέτρο. Διότι έχουμε ύψιστα ποσοστά και εντυπωσιακά ποσοστά ασφαλεία στην Ευρώπη. Ας μην ε, σπεύσουμε λοιπόν ε, με υπερβολική σπουδή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίτσεστερ. Και τώρα εκ μέρους της ε, Νοτικής Αριστεράς, για ένα λεπτό, η κυρία Βίλς. Σας ευχαριστώ. Στην Γερμανία προ λίγων ημερών 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της πυρηνικής ενέργειας και υπέρ των ανανεώσιμων ενεργειών. Και αυτά είναι δυνατόν να γίνουν. Μετά από το Τσερνομπίλ και το Φοκουσίμα είναι σαφές ότι πάντοτε θα υπάρχει κίνδυνος που θα ξεπηδά από τα πυρηνικά εργοστάσια. Γι' αυτό τα επίπεδα πυρηνικής ασφάλειας πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα υψηλότερα παγκόσμια επίπεδα και να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως σύμφωνα με το έγγραφο του Συμβουλίου του 2009 ισχύει μόνο το υψηλότερο επίπεδο ανά πάσα χώρα μέλος, αυτό που ισχύει στην νομοθεσία της δηλαδή. Χρειαζόμαστε τώρα νέα νομοθεσία με συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι στην βάση της συνθήκης Ευρατόμ. Εγώ τάσομαι υπέρ μιας πρωτοβουλίας των δυνατόν περισσότερων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να απευθύνεται στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επιτρέπει την ε, υιοθέτηση ενός χρονοδιαγράμματος αποχής από την πυρηνική ενέργεια. Για την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, για ένα λεπτό, η κυρία Τζαβέλα. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα και για το μορατόριο. Πρέπει να το σκεφτούμε αύριο. Αυτό που πρότεινε ο κύριος Τσίτσεστερ. Θέλω να προσθέσω ωστόσο τα εξή. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, ένα νέο κόσμο. Όλες οι φυσικές καταστροφές που θα εμφανιστούν τον 21ο αιώνα έχουν τεράστια μεγέθη, μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες, μεγάλα τσουνάμι. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε έναν πυρηνικό κίνδυνο λόγω των καταστροφών αυτών. Βλέπουμε ότι κινδυνεύουμε να φτάσουμε και σε τεράστιες ε, σε, σε φόνους σε μεγάλο αριθμό λόγω αυτών των καταστροφών. Κάνουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι η ΤΕΠΚΟ, η, αποτελεσμα... η έλλειψη αποτελεσματικότητας της ΤΕΠΚΟ είναι ένα νέο είδος εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Δεν έκανε, δεν έλαβε κανένα μέτρο, δεν πρόσεξε και θέλω να ζητήσω από όλους σας να σκεφτείτε αυτό το νέο έγκλημα, αυτά τα νέα εγκλήματα κατά της ε, κοινωνίας που θα αντιμετωπίσουμε τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ κύριε Τζαβέλα. Προχωρούμε στους υπόλοιπους αγορητές. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο η κυρία Ντελκαστήγιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να φάμε, για να ταξιδέψουμε, για να μελετήσουμε, για να θεραπεύσουμε ασθένειε. για πάρα πολλά πράγματα χρειαζόμαστε ενέργεια. Η ενέργεια αυτή πάντα προερχόταν από διάφορες πηγές. Σε κάποιες περιπτώσεις παλιότερα την υδροελεκτική, την ορυκτή και την πυρηνική. Όχι μόνο νέε όπως τι ανανεώσιμε. Υπάρχουν τεχνολογίες που εξελίσσονται επιπλέον για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ορισμένε περιπτώσεις. Υπάρχουν έρευνε ενέργειε που, ενέργειες που ερευνώνται και που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και που αυτή που φερειπίν αφορά την σχάση, την σύνδεξη, συγγνώμη. Αυτό, όλα αυτά εξελίχθηκαν κυρίε και κύριοι, βάση του ότι χρειάζεται να εξελισσόμαστε γιατί εξελίσσονται οι πόροι. Η έρευνα το πέτυχε αυτό. Ε, η επικοινωνία, η ιατρική, η μελέτη συνεχώς προσέβλεπαν στη βελτίωση των πόρων. Σήμερα το τσουνάμι και ο σεισμός οδήγησαν σε σοβαρότατες ε, βλάβες για την Ιαπωνία. Υπάρχουν θύματα, υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν υλικέ και μη υλικέ ζημιές. Υπάρχει μεγάλη ζημιά στον σταθμό της Φουκουσίμα. Καταρχάς ωστόσο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Αύριο θα ψηφίσουμε ένα κοινό ψηφισμά που συμφωνήσαμε η μεγάλη πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ομάδων και εκφράζει αυτό που μας ενώνει, όχι αυτό που μας χωρίζει. Ζητώ από τις ομάδες να είναι πιστοί στο περιεχόμενο της πρότασης και να μην βάλουν μπροστά τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους από τα κοινά συμφέροντα, από την κοινή άποψη που καταφέραμε στην πρόταση αυτή. Αυτή είναι η ευθύνη μας για αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντελκαστήλιο. Τον λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Ριέρα. Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη βαθιά λεγγύη με, τα, με τις οικογένειες των θυμάτων και με τα θύματα. Επίσης, τι δίδαγμα πρέπει να αντλήσουμε από αυτό το ατύχημα. Την επίγουσα ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα ασφάλειας. Η ασφάλεια ωστόσο περνάει και από τους ανθρώπινους πόρους. Χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο επίπεδο κατάρτισης για το προσωπικό που δουλεύει στον κλάδο. Χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι ότι οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικές. Κυρίες και κύριοι, η δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού και πλαισίου και πλαισίου κατάρτισης είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε ως ομάδα στο πρόγραμμά μας Ενέργειας για την Ευρώπη, που είναι μία έμφαση στα ανανεώσιμα, στις υποδομές, στην ενεργειακή απόδοση και την σύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για τον άνθρακα εφόσον είναι η μόνη εγχώρια πηγή ορυκτής ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ριέρα. Για ένα λεπτό η κυρία Χόλ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ε, δοκιμές αντοχής, τεστ αντοχής ε, δεν αρκούν να γίνονται με βάση κάποιες τεχνικές προδιαγραφές γιατί το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ο σεισμός το πρόβλημα στην Ιαπωνία ε, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η ανεπάρκεια της ενέργειας και, το, και η διατάραξη των συγκοινωνιών. Έτσι λοιπόν αυτό το ατύχημα στην Φουκοσίμα έχει, είναι πολυδιάστατο και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οι λοιποί ε, παράγοντε, οι λοιπέ συνθήκε που θα επέτρεπαν την αντιμετώπιση τη καταστροφή νωρίτερα. Και ε, δυστυχώ διαπιστώνεται ότι ακόμη συνεχίζεται η διαρροή ε, ραδιενεργά μολυσμένου νερού στι θάλασσε. Χρειάζονται λοιπόν και γεωμετρικές διαστάσεις στην καταμέτρηση αυτών των επιπτώσεων, όχι μόνο γεωλογικές μάλλον διαστάσεις, όχι μόνο τεχνικές. Ε, έχετε εσείς την ε, ευθύνη της πυρηνικής ασφάλειας, ε, κύριε Επίτροπε, έστω και αν λέτε ότι είναι απόφαση των κρατών μελών το αν θα σταματήσει η λειτουργία μιας πυρηνικής, ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι επενδυτές θα δώσουν περισσότερη έμφαση στο πόσο θα δεσμευτούν περισσότερο στην αποτελεσματικότητα της χρήσης ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές. Ευχαριστώ κύριε Χόλ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Τσουρμές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τραγικά περιστατικά της Ιαπωνίας μας δείχνουν πως το μόνο απόλυτα ασφαλές πυρηνικό εργοστάσιο είναι αυτό που δεν χτίστηκε ποτέ ή αυτό που έχει κλείσει είναι το μόνο απολύτω ασφαλέ πυρηνικό εργοστάσιο. Όλα τα άλλα αποδείχθηκε από την Ιαπωνία και μετά ότι είναι ε, ψέματα. Και το γνωρίζουν αυτό οι πολίτε Ευρώπη. Καθώ λοιπόν το γνωρίζουν οι πολίτε Ευρώπη, περιμένουν από εμά μια απερίφραστη και σαφή απάντηση. Η οποία απάντηση, η οποία ανταπόκριση πρέπει να είναι μόνο ότι η, ε, ο δικό μα οραματισμό στην Ευρώπη είναι η οικοδόμηση μέσων ανανεώσιμε πηγή ενέργεια με ε, ενεργειακά ε, οικονομικά σπίτια, με ενεργειακά ε, οικονομικές μεταφορές, με την μετάβαση μέσω του φυσικού αερίου από την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων στις ανανεώσιμες πηγές και εσείς κύριε Επίτροπε λέτε ότι πρόκειται να ετοιμάσετε τον οδικό χάρτη για το 2050, την ενέργεια στο 2050. Είσαστε διατεθειμένος λοιπόν να επεξεργαστείτε αυτό το όραμα μαζί μας, είστε πεπισμένος ότι αυτός ο ενεργειακός οδικός χάρτης θα έπρεπε να είναι ένας χάρτης ο οποίος όντως θα αξιοποιηθεί και ο οποίος όντως θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση και διάλογο με τον πολίτη της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τούρμες. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Ζημάνσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα διδάγματα, αν είναι να μάθουμε κάτι από τα γεγονότα στην Ιαπωνία, είναι να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Η πυρηνική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα της εξάρτησής μας. Βλέπουμε ότι στα σύνορά μας εμφανίζονται όλο και περισσότεροι πυρηνικοί σταθμοί που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε που δεν μπορούν να ελέγξουν οι νομοθέτες το νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις στο Καλίνιγκραντ, επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς και στο Καλίνιγκραντ και στην Λευκορωσία. Αυτό δεν θα είναι καλό νέο για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και της βιομηχανίας ενέργειας της Ένωσης προφανώς. Σήμερα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εκτός συνόρων θα υφίσταται, θα αντιμετωπίζει τα ίδια stress test όπως και η δική μας ενέργεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράμπστοφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταστροφή στην Ιαπωνία μπορεί να οδηγήσει σε έναν αριθμό συμπερασμάτων. Η ενέργεια θα πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του κράτους, υπό δημόσιο έλεγχο. Ή οσδήποτε σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να έχει και βοηθητικά συστήματα. Η ΤΕΠΚΟ απεδείχθη αμελής. Θα πρέπει να πούμε όχι σε αυτό το ξεπίδημα του φόβου που κυρίως προκαλούν οι δηλώσεις των πράσινων στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια επιτροπή ανθρώπων οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν νέες λύσεις, να έχουν πρωτοπόρο πνεύμα και να το αποδείξουν. Αυτό που δεν μας χρειάζεται είναι άνθρωποι οι οποίοι να εξετάζουν μοναχά τα προσωπικά τους, ατομικά τους συμφέροντα. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω το κοινό ψήφισμα με όλη μου την καρδιά. Αυτό δίνει ιδίω δύο μηνύματα στους αρμοδίους της χώρες μέλη αλλά και στο κοινό. Χρειαζόμαστε αφενός κοινού κανόνες για την προστασία από ατομικά ατυχήματα, πυρηνικά ατυχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οποιαδήποτε αμέλεια πρέπει να ανοίξει το παρελθόν. 180 χιλιόμετρα από το Στρασβούργο στη Γερμανία υπάρχουν δύο παλαιότερης τεχνολογίας πυρηνική σταθμή στη Γερμανία που ήδη υπολειτουργούν και άλλα, ε, και άλλα εργοστάσια έχουν κλείσει τελείω. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κοινά κριτήρια και τα χρειαζόμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχει η νομική βάση. Το ζήτημα είναι το ζήτημα πολιτική βούληση κατά πόσο θα προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι το έχουμε πράξει μέχρι τώρα. Δεύτερο, ό,τι και αν αποφασίσουν οι χώρε μέλη, ορισμένε χώρε μέλη θα αποσύρουν τα εργοστάσια από τη λειτουργία νωρίτερα, άλλε όχι. Αυτό όμως δεν πρέπει να αντισταθμιστεί με περαιτέρω αύξηση εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η στρατηγική 2020 δείχνει το σωστό δρόμο. Περισσότερες ανανεώσιμες ενέργειες, περισσότερη αποδοτικό, αποδοτικότητα της ενέργειας. Αυτά πρέπει να υλοποιηθούν κύριε Επίτροπε. Και εγώ συμπαρατάσσομαι με την πλειοψηφία του σώματος. Η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε τεράστιες εξοικονομήσεις. Και εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Ευχαριστώ. <clears throat> Για ένα λεπτό κυρία Τρότμαν. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανθρακική ενέργεια, αλλά μεταβατική ενέργεια. Και αυτή στηρίζεται σε εξαντλήσιμους πόρους και είναι ενδυνάμει επικίνδυνη. Η προτεραιότητα μετά τη φουκουσίνα είναι να δούμε την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών κατά βάση με συντονισμένο τρόπο σε επίπεδο ένωσης και να προχωρήσουμε να κοιτάξουμε και τι γίνεται κοντά μας ε, δουλεύοντας με απαιτητικούς κανόνες, με διαφάνεια και με ανεξάρτητους φορείς. Κατόπιν, η μάχη για την καταπολέμηση της αύξησης του κλίματος απαιτεί φιλόδοξη και συνεκτική πολιτική. Εάν με, την πυρηνική ενέργεια μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από αυτή την ενέργεια. Η Γαλλία παράγει ενέργεια από πυρηνικό σταθμό. Χρειάζεται να μειωθεί το ποσοστό της στο energy mix σαν προϋπόθεση. Για, ε, η έμφαση θα πρέπει να είναι εξοικονόμηση, αύξηση των ανανεώσιμων που θα έπρεπε να καλύπτει το σύνολο της κατανάλωσης. Μιλάμε για ασφάλεια πυρηνικών σταθμών. Θα πρέπει να μιλάμε επίσης και για ασφάλεια της τροφοδοσίας όλης της Ένωσης, ούτως ώστε καμία χώρα να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά την οικονομία της. Επίσης, να, μια πραγματική ελεγγύη σημαίνει να υπάρξει μια κοινότητα ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Τρότμαν. Για ένα λεπτό, η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ασφάλεια. Ναι, δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι για την ανεξαρτησία που είναι απαραίτητη ε, των αρμοδίων για την εξαγωγή των τεστ αντοχής και πρέπει οι προδιαγραφές να οριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ας μην ε, αυταπατώμεθα, έχουμε πεπαλαιωμένους πυρηνικούς σταθμούς που έχουν ε, κατασκευαστεί χωρί να λαμβάνονται υπόψη τέτοιου είδου υψηλή κίνδυνη. Άρα και με τεστ αντοχή και χωρί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατασκευάσουμε εγκατάσταση αντιδραστήρα πυρηνικό με βάση αυτού του παλιού, να του να μετατρέψουμε έτσι ώστε να είναι απολύτω ασφαλής. Αυτό δεν είναι ο κίνδυνο αυτό είναι ε, που δεν μπορούμε να τον ε, δεχθούμε για λογαριασμό του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα λοιπόν πρέπει και με τις οικονομικές δυνατότητες, οι ανάγκες και με την ανάγκη για απασχόληση και με, με, την, με το δεδομένο ότι πρέπει να αυξηθούν οι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα να χαράξουν μια πολιτική. Πώς θα γίνει αυτό με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο που θα σημαίνει Κλοντ είπε 15, στα, μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, ίσω είναι υπερβολικά αισιόδοξο, λίγο περισσότερο μπορεί να πάρει. Που θα σημαίνει λοιπόν ότι θα εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια και έτσι θα ξανακερδίσουμε τον πολίτη, την εμπιστοσύνη στου εαυτού μα, αλλά και στα θεσμικά όργανα. Γιατί πίσω από τη Φουκοσίμα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε να κάνουμε, υποκρύπτεται ένα, μία πράξη και παραγνώριση τη κρατική εξουσία και των αρχών εποπτεία. Αγνοήθηκαν αυτέ, με αυτό έχουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Τσχοτσμάν. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει ζητήσει να θέσει μια ερώτηση με το μπλε δελτίο. Συμφωνείτε. Μάλιστα, κύριε Ρούμπιχ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ να παρακαλέσω την κυρία Τροτμάν να μου πει στην Γαλλία υπάρχει το μοντέλο των ανεξάρτητων εποπτών που λειτουργεί πολύ καλά. Θεωρείτε ότι αυτό το γαλλικό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί συνολικά στην Ευρώπη για να υπάρξει ένας Ευρωπαίος ρυθμιστής σύμφωνα όπως είπαμε το γαλλικό πρότυπο. Ευχαριστώ τον κύριο Ρούμπικ που έθεσε την ερώτηση αυτή. Όντω, η γαλλική ρυθμιστική αρχή είναι ανεξάρτητη. Στη λογική αυτών που είπα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέργεια, θα έπρεπε να υπάρχει ένας, μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο με επαρκείς δυνατότητε ελέγχου με ανεξαρτησία και να μπορεί να υλοποιήσει το έργο της πραγματικά με ανεξαρτησία. Θέλετε να θέσετε ερώτηση σε συμπατριώτη στη σας κυρία Τρότμαν. Για την κυρία Τρότμαν λέει η κυρία Λεπάζ. Είναι ανεξάρτητη τυπικά η αρχή αλλά λόγω της σύνθεσης που περιλαμβάνει και του ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός μεταξύ αυτών πολλά ερωτήματα μπορούν να τεθούν ως προς την πραγματική της ανεξαρτησία. Κύριε Πρόεδρε, πάντα σε εθνικό επίπεδο μπορεί να αμφισβητεί κάποιο τη σύνθεση τη επιτροπή αυτή. και συμφωνώ επ' αυτού με την κυρία Λεπάζ. Πιστεύω ότι σύντομα θα περάσουμε σε μια περίοδο κατά την οποία θα μπορέσει να εξασφαλιστεί περισσότερο ο πλουραλισμό, Δεν θέλω ωστόσο να αμφισβητήσω την εντυμότητα της δουλειά των ατόμων που ανέλαβαν σοβαρά τι ευθύνε του, του κύριου Λακώστ ιδιαίτερα. Όλοι είναι ικανοποιημένοι. Να συνεχίσουμε. Κύριε Τρότμαν, βεβαίω. Ζήτω η Γαλλία, βεβαίω. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Τοσενόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ και μερικές εβδομάδες παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα γεγονότα που ακολούθησαν ε, τον ε, καταστροφικό σεισμό και το παλαιριακό κύμα στην Ιαπωνία. Θα ήθελα να σημειώσω το θαυμασμό που τρέφω για τους Ιάπωνες για τον τρόπο που διαχειρίζονται την κατάσταση αυτή. Τέτοιου είδους καταστροφές, καταστάσεις πολλές φορές ε, συνοδεύονται από πρόσθετα μέτρα. Μετά ένα πυρηνικό αεροπορικό δυστύχημα Φερρυπίνη, εισάγονται νέα μέτρα ασφαλείας για τις αερομεταφορές. Η καταστροφή λοιπόν στη Φουκουσίμα θα πρέπει να μας οδηγήσει στη δημιουργία νέων μέτρων, στην πρόβλεψη νέων μέτρων και αυτά τα τεστ αντοχής θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην υιοθέτηση των πλέον αυστηρών προδιαγραφών τα πυρηνικά εργοστάσια θα πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν στις πιο ακραίες συνθήκες και αυτό με βάση και τα όσα έχουμε δει στην ιστορία μέχρι τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν απλές και λογικές λύσεις γιατί είναι πολύ αυτονόητο, πολύ λογικό να ζητά κανείς να γίνεται δοχής στα πυρηνικά εργοστάσια. Τα γεγονότα της Ιαπωνίας αποτελούν μια ευκαιρία, χωρίς πολιτικές εταιρείε να ζητήσουμε την ε, επανεξέταση της αντοχής αυτών των πυρηνικών εργοστάσεων. Ευχαριστώ κύριο Ροήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ο καθένα γνωρίζει ότι στι χώρε μέλη, αλλά και εδώ μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν πολύ διαφορετικέ απόψει σχετικά με την χρήση τη πυρηνική ενέργεια. Και στην σημερινή συζήτηση διαπιστώνω ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει και μέσα στι πολιτικέ ομάδε. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, μια καταστροφή στην Ιαπωνία. Και αρχίσαμε μια συζήτηση και νομίζω ότι το ψήφισμα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία ώστε όλοι να εγκύψουμε σε ένα ερώτημα σήμερα και αύριο. Μπορούμε μαζί να ανυψώσουμε τα επίπεδα ασφαλείας και να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή κοινο, μια, ένα ευρωπαϊκό κοινό στοιχείο, μια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Ορισμένα δεν μου αρέσουν στο ψήφισμα. Όμως αυτό που κατόρθωσαν οι συνάδελφοι είναι μεγαλειώδες, ότι έφτιαξαν δηλαδή ένα κείμενο το οποίο περιορίζεται ε, ρίχνει το ιδιαίτερο βάρος του στα κοινά στοιχεία. Και διαρωτώ με αν δεν θα ήταν μια ευκαιρία σήμερα και αύριο να αφήσουμε λίγο στην άκρη το ερώτημα ναι ή όχι πριν εργοστάσια. Ας το αφήσουμε για λίγο εκτός παρενθέσεως και να ρίξουμε ιδιαίτερα το βάρος μας σε αυτά που είπα. Εάν δεν καταθέσουμε υποθετικά, εάν δεν ψηφίσουμε τις τροπολογίες μας αύριο και κατορθώσουμε να ψηφίσουμε ίσως και ομόφωνα ότι θέλουμε ασφάλεια και ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Τότε θα έχουμε προσφέρει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κύρος του, αλλά και στο ίδιο το θέμα, ποια συμπεράσματα δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε από την καταστροφή της Ιαπωνίας, μια μεγάλη υπηρεσία. Την συζήτηση ναι ή όχι πυρηνική ενέργεια μπορούμε να την κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να το σκεφτείτε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ, ε, συγγνώμη. ορίστε παρακαλώ. Τι απόγευμα είναι αυτό. Δέχεστε, Δέχεστε ερώτηση από την κυρία Χάρμς, κύριε Ρόιλ. Κύριε Ρόιλ, ε, γνωρίζετε ότι δεν είμαι πάντοτε υπέρ των προσεγγίσεων της ασφαλείας ε, για την πυρηνική ενέργεια όπως έχουν συζητηθεί μέχρι εδώ. Η μεγάλη πλειοψηφία του σώματος προ δύο ετών ήταν κατά των ύψιστων προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουμε και ένα πρόσθετο μεγάλο πρόβλημα, αν αρχίσουμε τώρα να μιλούμε για νέα κοινή εμπιστοσύνη. Το Κοινοβούλιο δεν έχει στην ουσία απολύτως τίποτε να πει σε ολόκληρη αυτή την αντιπαράθεση. Οι αποφάσεις για την πυρηνική ασφάλεια και τις δοκιμασίες αντοχής γίνονται το πολύ πολύ στο Συμβούλιο και στην Ευρατόμ και το Κοινοβούλιο παραμένει εκτός των θυρών. Το πολύ που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας. Αν αυτή θα έχει κάποιες ε, αν θα μπορέσει να ασκήσει κάποια επιρροή ή όχι, αυτό είναι γραμμένο στα άστρα. Όταν λέτε εσείς τώρα ότι μπορούμε να αντιβούμε την παλαιά συνθήκη Ευρατόμ και να διασφαλίσουμε διαφάνεια σε όλους τους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας, τότε ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε κύριε Ρόελ. Η ερώτηση. Ο κύριος Ρόελ. Δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση, διότι βεβαίως δεν υπήρχε ερώτηση στην ε, παρέμβαση τη Αλλά δεν πειράζει. Εγώ προσπάθησα και θα εξακολουθήσω να προσπαθώ να ε, συμβάλλω ώστε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία. Βεβαίω γνωρίζετε ότι έχουμε εσεί και εγώ τελείω διαφορετικέ απόψει, τελείω αντίθετε απόψει. Κύριε Σουλτ, α προσπαθήσουμε να μείνουμε σοβαροί. Κυρία Χάρμ, νομίζω θα ήταν ένα τεράστιο μήνυμα ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων εάν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ περισσότερη ασφάλεια και υπάρχουν πολλά σχετικά μέσα στο ψήφισμα και πολλά και σημαντικά και πολύ περισσότερα από όσα έχουμε μέχρι τώρα αποφασίσει και πολύ περισσότερα από όσα μπορούσα εγώ να συμφωνήσω μέχρι τώρα. Έχετε δίκιο. Αν όμω κατορθώσουμε να βάλουμε περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη Ευρώπη, τότε μπορεί αυτό να σημάνει ένα μήνυμα και προ τι χώρε μέλη. Εάν προχωρήσουμε σε διαφωνίες αύριο, διότι βεβαίως έχουμε διαφορετικές απόψεις σχετικά με την εγκατάλειψη ή μη της ενέργειας, δεν θα έχουμε κανένα σπουδαίο μήνυμα να δώσουμε. Αυτό λέω εγώ όλο και όλο. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Διαδικαστικό από πλευρά του κ. Τσίτσεστερ. Πρόεδρε, πραγματικά αισθάνομαι προσβεβλημένος που η κυρία Χάρμς απλά με ξεφώνησε εκτός μικροφώνου, ενώ για τον συνάδελφο ζήτησε μπλε, μπλε κάρτα. Μήπως θα μπορούσε να έχω μια ισότιμη αντιμετώπιση από πλευρά τη. Κύριε Ρόιλ, ξανά, για τον κύριο Ρόιλ θέλετε ερώτηση. Ναι, δέχεστε και άλλη ερώτηση κύριε Ρόιλ. Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Ρόιλ, εάν έχει αλλάξει τίποτα στην δική σας προσωπική θέση. Το πουλόβερ που φορώ τώρα έχει ηλικία 30 ετών από τότε που κατεβαίναμε και διαδηλώναμε. Και μα είχαν πει και τότε οι εμπειρογνώμονε ότι ο κίνητο υπάρχει μία φορά ανά 10.000 έτη. Τώρα ωστόσο ο πρόεδρο του Ινστιτούτου Πότσταμ λέει 10.000 χρόνια. 400 όμω εργοστάσια ολόκληρο το χρόνο είναι κάθε 25 χρόνια. Κάθε 25 χρόνια συμβαίνει όμω ένα τέτοιο μεγάλο πυρηνικό ατύχημα. Πρώτα Τσερνόμπιλ, τώρα Φουκουσίμα. Αλλάξατε τη θέση σας λοιπόν στα θέματα αυτά. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι ασφαλή ή πιστεύετε κι εσείς ότι το μη δημιουργηθέν εργοστάσιο είναι αυτό που είναι το ασφαλέστερο. Κύριε Ρόιλ, έχετε μόνο 30 δευτερόλεπτα, μην το ξεχνάτε. Πώς ο ερωτών έχει πάντα τόσο περισσότερο χρόνο. Δεν είναι τόσο δίκαιο, ο κανονισμός. Η άποψη μου βεβαίως έχει αλλάξει, όχι όμως επί του ουσιώδους. Είναι άσχημο να μπορεί να κανείς να διατηρήσει τη γνώμη του. Την έχω όμως αλλάξει πολύ τη γνώμη μου. Δήλωσα προηγουμένως ότι συμφωνώ με το ψήφισμα εφόσον παραμείνει ως έχει. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή σε σχέση με παλαιότερα. Αυτό μπορεί να σας αρκεί ή μπορεί να μην σας αρκεί. Αλλά αυτό είπα και εγώ εμένω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε ομόφωνα το ψήφισμα αυτό. Λίγο ξεκουραστείτε τώρα και συνεχίζουμε. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κ. Λάινεν. Ακούσατε τον πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, τώρα θα μιλήσω εγώ ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι απόψεις μας βέβαια διαφέρουν. Η ύψιστη ασφάλεια για όλα τα πυρηνικά εργοστάσια νομίζω ότι είναι αυτονόητη και οι δικές σας δοκιμασίες αντοχής είναι το πρώτο βήμα κύριε Τίνκερ, αλλά δεν αρκούν. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και που να πάει πολύ βαθύτερα και να είναι πολύ θεμελιωδέστερη. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε εκτός από την ύψιστη ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε και ένα σενάριο αποχώρησης από την πυρηνική ενέργεια διότι πρόκειται για ενδεχόμενους κινδύνους που δεν μπορούμε να λάβουμε την ευθύνη τους. Κύριε Ρόιλ, και εσείς και οι άλλοι, οι φίλοι σας στο Βερολίνο έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι εσείς εδώ στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες, στο Στασβούργο ή στι Εσείς εμένετε στις δικές σας απόψεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μας δοθεί μια διατύπωση, ένα σενάριο, μια στρατηγική εγκατάλειψη πυρηνικής ενέργειας. Και αυτή την ευκαιρία την έχετε με τον δικό σας χάρτη του Ιουλίου φέτος 2011 κύριε Επίτροπε. Να, να μας δείξετε με ποιον τρόπο μπορούμε να φύγουμε πλέον από την πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ κύριε Λάινεν. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Καντσάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, σήμερα θέλω να αποτίσω φόρο τιμή σε όλα τα θύματα τη καταστροφή, πραγματικής καταστροφής στην Ιαπωνία. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, τόσο ανησυχή, ανησυχητική που θεωρώ, αλλά θεωρώ ότι πολιτική δεν είναι να κάνουμε επιλογές σε συνθήκες πανικού, να μείνουμε πάντα ορθολογικοί, να αντιμετωπίζουμε σωστά την πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η βάση είναι σημαντική για να προχωρήσουμε, γιατί ξεκινώντας από δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ένας είναι ουρανός, αλλά η γη μοιράζεται με, σε σύνορα που δεν έχει να κάνει τίποτα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεύτερη παρατήρηση. Εμείς πρέπει να προσ, προσβλέπουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που δεν έχει μία διάσταση. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει τρεις παραμέτρους που πρέπει να συνυπάρχουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Αν δεν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, θα πάμε, δεν θα πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Το ψήφισμα που υποβλήθηκε και με το οποίο είμαι απόλυτα σύμφωνος, και που έλαβε και μια ευρύτατη συνένεση από ό,τι φαίνεται, φτάνει στη σωστή στιγμή για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στον τομέα της ασφάλειας, στον, στο check-up, στον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πώς θα γίνει αυτό. Σεβόμενοι τις παραμέτρους που έχουμε τη δεσμευτεί να τηρούμε και υιοθετώντα αποφάσεις προς την κατεύθυνση της ανανέωσης και της ε, αποτελεσματικότητας. Λαμβάνοντας ωστόσο πόψη ταυτόχρονα ότι χωρίς να προχωρήσουμε στην κουλτούρα της καινοτομία στο ζήτημα αυτό και στην πορεία προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνουμε λάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καντσιάν. Ενημερώθηκε η Προεδρία ότι σήμερα είναι τα του κύριου Λάινεν. Χρόνια πολλά κύριε Λάινεν. Για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Χέρτσοκ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πυρηνική ασφάλεια πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα ανθρώπινο πρόσωπο. Πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του συστήματος όταν πρόκειται για κλείσιμο των ε, μονάδων, όταν πρόκειται για εισαγωγή μέτρων, ασφαλής κλπ. Όλα αυτά έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Άρα πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση και πιο καλές γνώσεις του πώς λειτουργεί η πυρηνική ενέργεια. Είναι απαραίτητο αυτό και για τη λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου και για την λήψη μιας απόφασης περί κλεισίματος του. Συμφωνώ λοιπόν ε, στην ιδέα της εξαγωγής τεστ αντοχής και συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε νέα στοιχεία στην οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Επίσης οι υπερσυνοριακοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται έστω και με μόνο στόχο να καθησυχάσουμε την κοινή γνώμη. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε οι εθνικές αρχές να είναι σε θέση να λάβουν δράση όπου χρειάζεται και να μπορούμε και εμείς να επέμπουμε και συμφωνώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από όλα τα πυρηνικά απόβλητα που έχουμε δημιουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Πάνω απ' όλα πρέπει να μεριμνούμε για τους 500.000 πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Φράνκο, Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η βελτίωση πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να είναι το θέμα μα σήμερα. Όχι η αμφισβήτηση τη πυρηνική ενέργεια ως ε, των πυρηνικών ως πηγής ενέργειας για μη εισαρωτικούς ε, σκοπούς και της αποτελεσματικότητας της χρήσης αυτής. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν πρωτοβουλία για τα τεστ αντοχής στο σύνολο των πυρηνικών μας εγκαταστάσεων είναι ένα πρώτο και απαραίτητο βήμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να δεξαχθούν αυτά τα τεστ αντοχής με βάση μια κοινή προσέγγιση, με κριτήρια κοινά, με μεθοδολογία την οποία θα πρέπει να χαράξει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρχών Εποπτείας. Τα δε όμορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα πρέπει επίσης να υποβληθούν στις ίδιες δοκιμές αντοχής σε σχέση με τους κινδύνους ενδεχομένως μόλις περάσουν των συνόρων. Πέραν αυτών των τεστατοχή όμω, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει τα ύψιστα δυνατά στάνταρ, τι ύψιστα δυνατέ προδιαγραφέ σε διεθνέ επίπεδο για την πυρηνική ασφάλεια. Στο πλαίσιο τη G20, τη ομάδα των 20, τη Διεθνού ε, Υπηρεσία Πυρηνική Ασφάλεια και για την ε, ανάπτυξη των αντιδραστήρων. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνουμε και να προαγάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτεία τη πυρηνική ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει πρότυπο. Είτε πρόκειται για, για εφαρμογή κανονών, είτε πρόκειται για επίδειξη ελεγγύης, πρέπει να είμαστε το πρότυπο. Έναντι μια τέτοια τραγωδία, η δημιουργία μια αρχή πολιτική προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, πιστεύω, αδύρυτο ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό το λόγο θα λάβει τώρα η κυρία Φανμπρέμπτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η συνένεση για την πυρηνική ενέργεια ή η αντιπαράθεση με την πυρηνική ενέργεια μέσω των... είναι κάτι εγκάρσιο σε όλες τις ομάδες. Μετά τη Φουκουσίνωμα, ωστόσο, ξέρουμε ότι τέτοιες καταστροφές είναι πιθανές και σε εμά. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τρεις φάσεις. Πρώτον, τα stress test τα σχολεία, τα σχολεία και ο Επίτροπος πρέπει να προχωρήσουν με διαφάνεια. Πρέπει ωστόσο να έχουν και συνέπειες. Εάν μια, ένας σταθμό σταθμός δεν είναι ασφαλής, κλείνει. Δεύτερη φάση, να οργανώσουμε ένα phasing out της πυρηνικής ενέργειας. Είναι απαράδεκτο ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτίστηκαν με 20-30 χρόνια διάρκεια ζωής να λειτουργούν μετά από 40 ή 50. Τρίτον, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και τη δουλειά μας στις ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαμπρέμπτ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Σόνικ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στις 26 Απριλίου θα πέρασε θα έχουμε 25 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ. Καιρός είναι να θυμηθούμε κι εμείς λίγο τα θύματα του ατυχήματος αυτού. Ταυτόχρονα θυμάμαι τις εξελίξεις, την κατάσταση τότε στο Τσερνομπίλ και θέλω να εκφράσω την κατανόησή μου και την ε, και τη συμπαράστασή μου στο λαό της Ιαπωνίας που αγωνίζεται και αυτός με ε, μια πυρηνική ενδυνάμει καταστροφή. Ο Κέσιο 137 έχει ζωή 30 ε, ετών και μπορεί να ε, επηρεάσει όλα τα είδη που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η Greenpeace μιλάει ότι η μόλυνση αυτή μπορεί να περάσει από το ένα προϊόν στο άλλο. Η δε περιοχή ε, μόλυνσης έφτασε σε ανώτατα επίπεδα ε, σε μία, περίμετρο 30, χιλιόμετρων γύρω από το Τσερνομπίλ. Η Ευρώπη έχει στα σύνορά της σοβαρούς κινδύνους και η Λευκορωσία και η Ρωσία χτίζουν νέους πυρηνικούς σταθμούς των οποίων τα πυρηνικά τα, στάντα δεν γνωρίζουμε. Όποια και στάντα να υιοθετήσουμε και όποια stress να υιοθετήσουμε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή την κατάσταση. Ε, ε, ίσως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο ε, πιο, όχι τόσο γρήγορα κύριε Σόνικ, θα μπορούσατε. Ξαναλέω αυτά που έλεγα πρόεδρε. Η Ρωσία και η Λευκορωσία χτίζουν τώρα πυρηνικούς σταθμούς δίπλα στα σύνορα της Ένωσης. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα έπρεπε να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμού τέτοιου που δεν μπορούν να περάσουν τα ίδια στρες τεστ όπως η Ευρωπαϊκή Πυρηνική Σταθμή. Ο κύριος Έντσιο, ένα λεπτό. Πρόεδρε, θέλω καταρχά να εκφράσω την τα συλληπιτήριά μου και την πλήρη συμπαράστασή μου προς το λαό της Ιαπωνίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε πραγματικά. Το ατύχημα της Φουκουσίμα δείχνει ότι κανένας πυρηνικό σταθμό δεν είναι απόλυτα ασφαλή. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα πυρηνική ασφάλειας και να προωθήσουμε το συντομότερο δυνατό κείμενα για την ασφάλεια των σταθμών αυτών. Επιπλέον, δεν πρέπει, από την πλευρά, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα των αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση συναισθηματικές ή βεβαιασμένες ε, σκέψεις. την απόφαση ε, εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας. Τα πρώτη μέρη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα το ενεργειακό τους μίξ υπό τον όρο βεβαίως ότι θα τηρούν τα ίδια στάνταρ ασφάλειας. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται και σε έναν υψηλό βαθμό επιστημονικής γνώσης. Ο κύριος Καρίνης έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Αξιότιμα Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η πυρηνική ενέργεια εξασφαλίζει τώρα περίπου τρίτο τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο στην Ευρώπη. Εάν θέλουμε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντικαταστήσουμε αυτή την πηγή, θα πρέπει να έχουμε δύο, έχουμε δύο εναλλακτικέ. Δηλαδή, είτε θα πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση του ε, άνθρακα, είτε αυτήν του φυσικού αερίου. Και οι δύο όμως αυτές εναλλακτικέ έχουν σημαντικά μειονεκτήματα. Παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα ε, για το κάρβουνο και προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία κυρίως για το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση και νομίζω ότι αυτή είναι η ενίσχυση της ασφάλειας. Ωστόσο αγαπητοί συνάδελφοι δεν αρκεί να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας μόνο στην Ευρώπη διότι ε, στα σύνορά μας ε, γύρω από την Ευρώπη τη Ρωσία συγκεκριμένα και τη Λευκορωσία ε, έχουμε αντιδραστήρες οι οποίοι προχωρούν ε, χωρίς να γίνονται σεβαστές οι προδιαγραφές ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν ύψε προδιαγραφές ασφαλείας να ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στα κοντινά κράτη όπω η Ρωσία και η Λευκορωσία. Και δεύτερον, μπορούμε στην Ευρώπη να ενισχύσουμε μέτρα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας και να χρησιμοποιούμε άλλες εναλλακτικές ενέργειες όπως την υδροηλεκτρική, την ηλιακή, το, τα βιοκαύσιμα και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα μπορούμε να εισαγάγουμε μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια όπω έλεγα. Η αιωλική, η ηλιακή ενέργεια, η βιομάζα μπορούν να μα επιτρέψουν να απεμπλακούμε περισσότερο από την πυρηνική ενέργεια αλλά και από τι αγωγέ άλλων καυσίμων. Ευχαριστώ. Ο κ. Σπυρίλο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πληροφορίε από τη Φουκουσίμα είναι όλο και πιο ανησυχητικέ. Ξεπεράστηκαν κατά πολύ τα όρια ασφάλεια, Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο εγγύς μέλλον δεν υπήρξε σαφής επικοινωνία ούτε διαφάνεια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στα στρες τεστ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αν υπάρξουν προβλήματα στην έκβασή τους θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ζητήσουμε την άμεση διακοπή λειτουργίας των σταθμών αυτών πρέπει να τηρούμε τις υψηλότερες δυνατές παραμέτρους ασφάλειας και να μην προχωρήσουμε σε κατασκευή νέων σταθμών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ε, σταδιακή διακοπή χρησιμοποίησης ενέργειας αυτής που μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε στο μέλλον πολιτικές ενέργειες που θα που θα στοχεύουν στην αποταμίευση ενέργειας, στην απόδοση και να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εν τέλει θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση στην οποία θα μετέχουν και οι πολίτες και η τοπική διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πυρίλο. Για 1,5 λεπτό, λεπτό η κυρία Γιόνταν. Πρόεδρε, συμφωνώ με εκείνου συναδέλφου οι οποίοι είπαν ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πυρηνική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κουλτούρα περί ασφάλεια είναι ευρύτατη έννοια. Σημαίνει και ασφαλή πυρηνική τεχνολογία, αλλά και διασφάλιση τη κατάλληλη χρηματοδότηση των πόρων, δηλαδή ανθρωπίνων και υλικών, ε, των προδιαγραφών ασφαλεία και μια ανεξάρτητη ε, εποπτική αρχή. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν μιλούμε για τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ ασφαλεία. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν σεβόμαστε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη καλύτερα στου φυστόμενου θεσμού και τα όργανα που υπάρχουν ήδη, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και σε θεσμικό επίπεδο τι υψηλέ δυνατέ προδιαγραφέ. Είπατε εσεί μάλιστα κύριε ότι τα κράτη-μέλη δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Στην τελευταία ανάλυση όμω θα ρωτήσουμε ποια είναι τα κράτη-μέλη. Εάν ρωτήσουμε τον πολίτη μα, εάν ρωτήσουμε την κοινή γνώμη, και έχουν γίνει σχετικέ δημοσκοπήσει. Εάν ρωτήσουμε λοιπόν το, την κοινή γνώμη τι γίνεται, ε, τι γνώμη έχει, πιστεύω θα μα πει πω ε, θέλει να υπάρξει απαραίτητη ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά από την άλλη, για πολιτικού λόγου, καλό θα είναι να μην κλείνουν τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ιαπωνία. Πολλά είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Ένα μόνος μόνο όμω έχει πληγεί από αυτή την ε, τραγωδία, από το ατύχημα. Πριν λοιπόν να καταλήξουμε σε επιβεβαιασμένα μέτρα, καλό θα ήταν να έχουμε εμπεριστατωμένα στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία, μια επιστημονική ανάλυση που θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στη Φουκοσίμα για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος ή οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν στο πυρηνικό ατύχημα και ε, τη ζημία στον ε, πυρήνα στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Τώρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των πυρηνικών αποβλήτων. Είμαστε έτοιμοι πιστεύω να δείξουμε ότι έχουμε με σοβαρότητα αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η κυρία Αλφάνο έχει σηκώσει μια μπλε κάρτα. Συμφωνείτε, δέχεστε την ερώτηση. Κύριε Αλφάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ζητήσω από τη συνάδελφο. Χιλιάδες νεκροί δεν είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να μελετήσουμε επί μακρόν. Ε, δεν έχουμε στοιχεία που να μας οδηγούν, είπε η συνάδελφος ότι δεν έχουμε στοιχεία που να μας οδηγούν ότι η πυρηνική σταθμή είναι επικίνδυνη. Με τους χιλιάδες νεκρούς στην Ιαπωνία αυτό δεν είναι ένα στοιχείο. Να το σκεφτούμε περισσότερο. Η κυρία Μέρκης. Μία ερώτηση. Πόσες, πόσοι πυρηνικοί σταθμοί πρέπει να κλείσουν γιατί είπατε για να είναι αρκετοί. Είπα, μιλήσατε για έναν. Για ένα πυρηνικό. Είπατε ότι ένας μόνο πυρηνικό σταθμός επλήγει. Δεν ήταν ένας. Έξι ήταν καταρχάς. Πόσοι είναι αρκετοί, για, πόσοι πρέπει να υπάρξουν για να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη. Ευχαριστώ. Come on. Ε, Προβλέπω ε. ότι θα μείνουμε πολύ αργά απόψε. Uh, Πρόεδρε, αν μπορούσα με τη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΕΑ να θέσω και εγώ ένα ερώτημα τώρα. Υπάρχει ένα περιοδικό εργοστάσιο και στη χώρα σας, το Κρίσκε, το οποίο αντιμετωπίζει ενδεχόμενα κίνδυνο διότι βρίσκεται στη σεισμογενή περιοχή. Θα είστε, θα είστε υπέρ της ιδέας να είναι από τα πρώτα εργοστάσια που θα κριθούν με τις δοκιμασίες αντοχής που ελπίζουμε θα είναι αυστηρές και αντικειμενικές ώστε να έχουν την πεποίθηση οι πολίτες ότι παρόλο που βρίσκεται στη σεισμογενή περιοχή το εργοστάσιο αυτό δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ή εν πάση περιπτώσει ότι μπορεί να βελτιωθεί όσο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Η κυρία ε, Να σας ευχαριστώ πρόεδρε. Στην Ιαπωνία, όντως, μετρήσαμε χιλιάδες θύματα. Προσωπικώς εκφράζω την οδύνη μου και τη συμπαραστασία μου. Πιστεύω ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να συμβάλλει στο βαθμό των δυναμεών της. Αλλά το να γίνεται κατάχρηση του αριθμού των θυμάτων για να αναπτυχθεί ένας πόλεμος κατά των πυρηνικών εργοστασίων, το βρίσκω υπερβολικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συστήσουμε τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτό το πυρηνικό ατύχημα και να δούμε αν είναι δυνατόν να εμφανιστεί αντίστοιχο πυρηνικό ατύχημα και στην Ευρώπη. Και δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα θύματα των φυσικών καταστροφών όπως ο σεισμός στο παλαιριακό κύμα με αυτά που μπορεί να προξενήσει ένα πυρηνικό ατύχημα. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Η δεύτερη ερώτηση. Πόσα, πόσα πυρηνικά εργοστάσια πρέπει να ε, δημιουργήσουν πρόβλημα, πόσα πυρηνικά ατυχήματα μου αρκούν. Σας είπα, ένα με πολλούς αντιδραστήρες. Ναι, ένα εργοστάσιο ήταν με πολλούς αντιδραστήρες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πυρηνικά εργοστάσια στην Ιαπωνία. Κάθε ένα από τα ατυχήματα πρέπει να εξετάζεται με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και όχι μόνο το ίδιο το ατύχημα, αλλά και όλες οι περιστάσεις που μπορεί να, ε, οι όλες οι συνθήκες, τα περιστατικά που μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ως ατυχήματα αλλά να διαβαθμίζονται διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ένα μόνο ατύχημα να οδηγήσει σε μια απόφαση βεβαιασμένη. Δεν έχω δώσει απάντηση σε ερωτήσεις μου πρόεδρε, ήταν τρεις ερωτήσεις που είχα. Μισό λεπτό ακόμη λέει ο πρόεδρος. Για δε το πυρηνικό εργοστάσιο στη χώρα μου. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με δοκιμή, με δοκιμή, ε, και οι Αυστριακοί έκαναν αντίστοιχες μελέτες για τη σεισμική ασφάλεια και κάποιες τροποποιήσεις στο εργοστάσιο του Κέσκο ε, ελήφθησαν τελικά. Σε αυτά συμφωνώ απολύτως και είμαι πεπισμένη ότι όλοι οι Σλοβαίνοι θα συμφωνήσουν πως πρέπει και στη Σλοβενία να πραγματοποιηθεί τεστ αντοχής. Είμαστε μικρό κράτος όμως σε πυρηνικού όρους και νομίζω ότι χρειαζόμαστε ίσως λιγότερους διεθνείς ελέγχους από ό,τι χώρες που έχουν περισσότερα εργοστάσια. Ο κύριος Ζίμπερ έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι Αυστριακός και η ανησυχία μας από το εργοστάσιο Κρέσκο μας ε, πλήττει όλους χαίρομαι και ελπίζω η υπόσχεση της συναδέλφου μου να ε, τηρηθεί. Η μεγάλη μου ανησυχία πάντως και συμπαράσταση πηγαίνει στον Ιαπωνικό λαό που με στοική υπομονή αντιμετωπίζει τα γεγονότα. Ας διδαχθούμε και κάτι θετικό από την κρίση και αυτό μπορεί να είναι ότι θα καθίσουμε να σκεφτούμε και εδώ στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε επιτέλους να συνάγουμε συμπεράσματα από την κρίση αυτή που βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι μόνον ότι πρέπει να αυξήσουμε σημαντικά τα επίπεδα ασφαλείας των ευρωπαϊκών αντιδραστήρων. Επίσης χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προστασία απέναντι σε θεομηνίες και καταστροφές. Μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Το δίδαγμα δεν μπορεί παρά να είναι να συντάξουμε όλοι μαζί σενάρια, χρονοδιαγράμματα εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας διότι υπό την παρούσα τουλάχιστον τεχνολογία δεν είναι δυνατόν να, ε, να απαλλαγεί κινδύνων η πυρηνική ενέργεια. Ούτε άλλωστε στο μέλλον πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπετε από την παρέμβασή μου ότι υπάρχουν πολλέ και ποικίλε απόψει και μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την πυρηνική ενέργεια. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένη. Γι' αυτό Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει με μονομένους κινδύνους. Δεν είχαμε μέχρι τώρα σωρευτικούς κινδύνους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό σενάριο. Πράγματα όπως ε, ένα παλιροϊκό κύμα τσουνάμι είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Αλλά σεισμογενείς περιοχές υπάρχουν και ασφαλώς ε, και εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μαρινέσκου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να εκφράσω τον θαυμασμό και το σεβασμό μου για τη στάση του Ιαπωνικού λαού ενώπιον αυτής της έκτακτης κατάσταση που αντιμετωπίζει. Κατόπιν, η συζήτησή μας αφορά το πυρηνικό μέλλον της Ευρώπης. Σταματάμε ή προχωράμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, λαμβάνοντα υπόψη τι πολλέ διαστάσει του προβλήματο. Ασφάλεια, κλίμα, ε, βούληση των πολιτών. Πρέπει να στηρίξουμε τη θέση μα σε ένα ενεργειακό μίξ. Ανανεώσιμε ενέργειε και παραδοσιακέ ενέργειε. Με ασφαλή τρόπο μεταξύ των οποίων και η πυρηνική ενέργεια. Θα πρέπει δε να προχωρήσουμε σε έρευνα, αποτελεσματική έρευνα στον τομέα των ανανεωτικών πηγών ενέργειας. Η έρευνα και η βελτίωση της τεχνολογίας θα πρέπει να μειώνουν και την ρήπαση των παραδοσιακών τεχνολογιών και την ε, βελτίωση των νέων μορφών ενέργειας. Πρέπει να βελτιώνουμε τις υφιστάμενες τεχνολογίες για να και τηρώντας αυστηρότερα στάνταρ. Τα stress test πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες κινδύνου. Φυσική κίνδυνη, αλλά και κίνδυνοι ανθρωπογενής. Θα πρέπει δε να γίνονται με συμμετοχή και της Επιτροπής. Τα τεστ δε πρέπει να δίνουν, να έχουν σαφή σκοπό. Όποιος περνάει το τεστ συνεχίζει, όποιος δεν περνάει κλείνει. Επιπλέον πρέπει να υιοθετήσουμε μια στρατηγική για την επεξεργασία και αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων και για το κλείσιμο κάποιων πυρηνικών σταθμών. Κάποιο, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι η κοινή γνώμη θα πρέπει να συνεχίσει να πιστεύει στην πυρηνική ενέργεια και να ενημερώνεται σχετικά. Λοιπόν, συνάδελφοι, 34 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο μέσω της διαδικασίας αυθόρμητων ομιλιών, catch the eye. Πολύ ζωντανή συζήτηση, πολλές μπλε κάρτες, ήμουν γενναιόδωρος στη διαχείριση του χρόνου. Λοιπόν, δεν θα δώσω το λόγο βέβαια σε 34 συναδέλφους. Κατ' εφαρμογή λοιπόν των αρμοδιοτήτων μου και με την άδειά σας, θα δώσω το λόγο δύο, σε δύο συναδέλφους από το ΕΛΚ, δύο στους σοσιαλιστές, έναν από τους Πρασίνους, ένα, έναν από τους φιλελεύθερους, έναν από τους Πράσινους, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος, έναν από το EFD και ένα στους μη εγγεγραμμένους. Η κυρία Αντρική έχει το λόγο. Ένα σχόλιο σύντομο για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε τρίτε χώρε κοντά στα σύνορα της Ένωσης. Δύο περιπτώσεις αναφέρθηκαν ήδη. Νέε εγκαταστάσεις, μία στο Καλίνιγκραντ, κομμάτι της Ρωσικής Ομοσπονδίας που περιβάλλεται απόλυτα από την Λιθουανία, την Πολωνία και την Βαλτική και ένα δεύτερο σταθμό στη Λευκορωσία, όπου προγραμματίζεται η κατασκευή ενός ε, πυρηνικού σταθμού 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Λιθουανίας. Όταν έβλεπε όλος ο κόσμος εξελίξει στη Φουκουσίμα, δραματικέ εξελίξει εκεί, η κυβέρνηση της Λευκορωσία στις 15 Μαρτίου και η Ράσατομ ρωσική ε, εταιρεία υπέγραψε μια συμφωνία για την κατασκευή νέου σταθμού στην Λευκορωσία το 2018. Επίσης η Ρωσία ετοιμάζει μια επένδυση για 6 δις δολαρίων στην Λευκορωσία για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού. Οι αρχές της χώρας δεν ενημέρωσαν επαρκώς τους, συναδέλφους, τους γείτονές της και κάτι τέτοιο παραβιάζει την σύμβαση του ΕΣΠΟ για, το, την μελέτη, για τις μελέτες περιβαλλοντικών δικτύπου. Ευχαριστώ. Η κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, Χαίρο για την απόφαση της Επιτροπής να υποβάλει σε stress τεστ τους πυρηνικούς σταθμούς της Ένωσης. Θέλουμε ο έλεγχος αυτός να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κοινών κριτηρίων, πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων για την περαιτέρω βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην Ένωση. Σήμερα, στο εσωτερικό της Ένωσης υπάρχουν πάνω από 130 πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στα, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνοι για το, το ενεργειακό τους μίξ. Ωστόσο η πυρηνική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Άρα πρέπει να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα για την πυρηνική ασφάλεια στο εσωτερικό της Ένωσης. Υπογραμμίζω ότι οι επενδύσεις στην ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών θα πρέπει να ισχύουν μέχρι τελευταία στιγμή λειτουργίας του κάθε σταθμού. Το στο μέλλον το κόστος της ενέργειας, από ενέργειας που παράγεται από πυρηνική ενέργεια θα αυξηθεί και θα έπρεπε να αναζητήσουμε ε, καλύτερη χρησιμοποίηση των ενανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κυρία Γιάτεν Μάκη έχει το λόγο τώρα. E Η Ένωση θέλει στα κράτη-μέλη και στις γειτονικές χώρες να γίνουν stress test. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικά. Η Ένωση ζητά ευγενικά να προχωρήσουν οι χώρες αυτές σε stress test. Άλλη δυναμία είναι ότι η Ένωση δεν έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες. Κάτι... Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Τρίτον, θα πρέπει να γίνουν τα τεστ τα από ανεξάρτητα όργανα. Δεν πιστεύω ότι οι εθνικέ ρυθμιστικέ ελεγκτικέ αρχέ θα πούν ότι στη δική του χώρα υπάρχουν προβλήματα ή αμέλεια σε επίπεδο ελέγχου. Θα, θα, θα πρέπει τα τεστ να είναι πραγματικά και να υπακούουν σε κανόνες ανεξάρτητους που τους διεξάγουν ανεξάρτητοι οργανισμοί. Η κυρία Ριβάζη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θέλω να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι δεν τελείωσε το ατύχημα της ε, Φουκουσίμα. Υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι εκρήξεων στο κέντρο του αντιδραστήρα. Μία ερώτηση προς τον κύριο Έτιγκερ. Η υλοποίηση των ε, stress test, είπε και ο συνάδελφος για το θέμα αυτό. Πώς θα φροντίσετε να είστε βέβαιοι ότι όλα τα κριτήρια που αναφέρετε στην Επιτροπή ΙΤΡΕ θα λαμβάνονται υπόψη από όλα τα κράτη που έχουν πυρηνικούς σταθμούς. Πώς θα υποχρεώσετε ένα κράτος που αρνείται να ελέγχουν ε, τους ε, σταθμούς ανεξάρτητοι ελεγκτές. Γιατί μεταξύ μας, αν οι ίδιοι είναι στον έλεγχο, πώς θα εφαρμόσουμε τα stress test. Θα πρέπει να είναι μια τελείως ανεξάρτητη δομή που θα κάνει τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σε όλα τα κράτη. Πώς θα φροντίσουμε οι γειτονικέ χώρες. Μιλήσατε για την Αρμενία, τη Λευκορωσία ακούστηκαν. Πώς θα τους πείσετε να δεχθούν κάτι τέτοιο. Θα πρέπει βεβαίω να σας υποστηρίξει το Κοινοβούλιο, αλλά τι θα κάνετε μετά. Για τις ευθύνες. Υπάρχει ευθύνη για να αυγούμε από την πυρηνική ενέργεια και πρέπει να προτείνουμε στο Κοινοβούλιο σενάρια αποχώρησης και εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας. Το μόνο, ο μόνος τρόπος για να μην έχουμε άλλα Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ. Οι ζημιές ε, στον αντιδραστήριο της Φουκουσίμα λόγω φυσικών καταστροφών δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να είμαστε βέβαιοι για την ασφάλεια τέτοιων εγκαταστάσεων. Γι' αυτό και καλά έκανε η Ένωση να προχωρήσει σε ελέγχους σε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς και καταστάσεις από ανεξάρτητους ε, ελεγκτές που θα δείξουν τους κινδύνους και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε. Είμαι βέβαιος ότι μετά την δημοσίευση των ευρημάτων του ελέγχου θα ληφθούν αποφάσεις που θα απαιτούν από τις επιχειρήσεις να περιορίσουν, να, να καταργήσουν τα και να, Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε ένας, ε, ένα εργοστάσιο να παρακάμψει, να καταστατηγήσει τα κριτήρια ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Κύριε Επίτροπε, το κοινό της Ευρώπης θέλει έναν ανοιχτό διάλογο για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη και μια αξιολόγηση όλων των σταθμών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία μας έδειξε ένα πράγμα. Η φύση είναι ισχυρότερη από τον άνθρωπο. Έχει έρθει η ώρα τα πυρηνικά εργοστάσια που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές να φύγουν από τα δίκτυα. Οι δοκιμασίες αντοχής, κύριε, ε, κύριε Επίτροπε. Όχι άλλο Τσερνόμπιλ. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εισαγωγές προϊόντων από την ε, Ιαπωνία. Θέλετε να μας ακτινοβολήσετε. Ας επενδύσουμε σε ε, ανανεώσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες. Υπάρχουν τέτοιες. Σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο και εκτός από αυτό δημιουργούν και απασχόληση. Στην Αυστρία είχαμε το εργοστάσιο Τσέμπτεντορφ το οποίο ποτέ δεν παρήγαγε πυρηνική ενέργεια και σήμερα παράγει ηλιακή ενέργεια. Ας επαναλάβουμε το παράδειγμα αυτό. Κύριε Μακίνης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά πήγε παραπέρα και μιλά για την, πυρηνική, για την πυρηνική ασφάλεια και ενώ μιλά για την πυρηνική ενέργεια. Η Επιτροπή θα έπρεπε να προχωρήσει έναν οδικό χάρτη για την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή. Σωστά χρησιμοποιούμε τον όρο stress test, γιατί στι τράπεζε δεν πήγαν καλά τα stress test. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε τον όρο αξιολόγηση εκτίμηση κινδύνου και να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι αξιολογήσεις θα γίνουν σε όλες τις εγκαταστάσεις ακόμα και αυτές που αφορούν την επανεπεξεργασία και ε, ανα, αναχρησιμοποίηση του υλικού. Φοβάμαι ιδιαίτερα για την κατάσταση στο Σέλαφιλτ. Πρέπει να δούμε την ασφάλεια των ε, υλικών. Λένε ότι εξαρτώμαστε πολύ από την πυρηνική ενέργεια παρότι δεν έχουμε επιτόπου ε, πυρηνικού σταθμού. Η ασφάλεια λοιπόν είναι καθοριστική. Ας δούμε ευρύτερα το θέμα του ενεργειακού μίξ και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δεν είναι εύκολη απάντηση οι ανανεώσιμε. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μα πήρε 25 χρόνια για να ξεχάσουμε το Τσερνομπίλ και φοβάμαι ότι η καταστροφή στην ιαπωνία δεν αρκεί για να μας το θυμίσει. κατηγορούμε συστηματικά την ιαπωνία. είναι σαν να θέλουμε να πούμε ότι είναι η ιαπωνία και όχι η πυρηνική ενέργεια που δεν ήταν ασφαλής. ξεκινάμε τεστ ασφαλείας για τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις και πάλι εμένουμε ότι υπάρχει ασφαλής πυρηνική τεχνολογία. χρειαζόμαστε να κλείσουμε άμεσα τι πυρηνικέ εγκαταστάσει άνω τριακονταετία και να σταματήσουμε κάθε σκέψη για κατασκευή καινούριων. χρειαζόμαστε άμεσα ένα φόρο πυρηνικών που θα μα επιτρέψει να απεικονίζουμε όλο το περιβαλλοντικό κόστο τη πυρηνική ενέργεια. πρέπει να επενδύσουμε στην αύξηση τη απόδοση των φωτοβολταϊκών και πραγματικά να επενδύσουμε στην αύξηση τη απόδοση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. επίτροπε εσεί έχετε την νομοθετική πρωτοβουλία και η ευθύνη της δράσης μας ή των επιπτώσεων της αδράνειας είναι και δική σας. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος κ. για έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, πρώτα για την μακροπρόθεσμη πολιτική ενέργειας. προσφέρω στις πολιτικές ομάδες ήδη από τον Μάιο να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην συζήτηση διαφόρων σεναρίων της διαχείρισης της ενέργειας για τις επόμενες δεκαετίες. Ένα σενάριο, δηλαδή μια επιλογή με όλες τις απαραίτητες επιπτώσεις θα σημαίνει βέβαια να είναι και υψηλό το ποσοστό των ανανεώσιμων ενεργειών με επιπτώσεις για τα δίκτυα, για την έρευνα, για τις δυνατότητες αποθήκευσης και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα θα παρακαλέσω να εξεταστεί και το νομικό πλαίσιο. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ζωή μονάχα 1,5 χρόνου. Και εσείς συμμετέσχατε περισσότερο από ότι εγώ στην διατύπωσή της. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ε, σημαντική νομοθετική αρμοδιότητα για το δίκαιο της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει μία, μία εξαίρεση, αλλά σημαντική και συνειδητά. Το ερώτημα της τεχνολογίας της ενέργειας, της energy mix, που είναι θέμα των εθνικών κοινοβουλίων. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε αν αυτό ήταν σωστό ή όχι, αλλά οι συνέπειες είναι σαφής. Και για τον οδικό χάρτη της ενέργειας, για να γίνει αυτός στην βάση της συνθήκης Λισαβόνας, θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να το ζητούμε. Ίσως είναι επιθυμητό. Και εγώ επιθυμώ, θεωρώ μάλιστα ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εμπειρογνωμοσύνη για θέματα ε, ενεργειακού μείγματος. Αλλά για τα επόμενα χρόνια πάντως είναι θέμα αρμοδιότητας των χώρων μελών. Ένας περιορισμός που είχαμε επιτύχει με τις χώρες μέλη, τα 20% δηλαδή των ανενώσιμων ενεργειών περιορίζουν στο 80% την αρμοδιότητα των χωρών μελών για την διαχείριση της ενέργειας είπαμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το 2020 τα 20% και αυτά θα τα εξετάζουμε και με εκθέσεις πρόοδου. Έτσι λοιπόν περιορίζεται η αρμοδιότητα των χωρών μελών στα θέματα ενέργειας στο 80% της ενέργειας αυτής. Και ακόμα λιγότερο. Γιατί? Διότι τα 20% ίσως σημαίνουν στον τομέα των μεταφορών 10%. Στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος που είναι σήμερα βέβαια στο επίκεντρο, μέσα στα επόμενα 9 χρόνια 35% των ανανεώσιμων ενεργειών, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, αιωλική ενέργεια, θα είναι 35%. Αυτό σημαίνει ότι σε 3 έως 4 χρόνια οι ανανεώσιμες ενέργειες θα έχουν ξεπεράσει τον άνθρακα και τα πυρηνικά εργοστάσια στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο. Βρίσκω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια διαδικασία εξέλιξης την οποία πρέπει να την εκτιμήσουμε ιδιαίτερα σε 9 χρόνια 35% ανανεώσιμες ενέργειες. Και με τον οδικό χάρτη της ενέργειας δεν θα βάλουμε μόνο ως ορίζοντα το 2050 αλλά και το 2025 για τα επόμενα χρόνια δηλαδή όπου χρειάζονται επενδύσεις και στα δίκτυα και στις, και στις ε, δυνατότητες αποθήκευσης. Άρα για να φτάσουμε στο 40% σύγχυ της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που όλο και περισσότερο περιορίζει το ποσοστό των χωρών μελών. Όταν οι ανώσιμες ενέργειες θα φτάσουν στο 40% τότε οι χώρες μέλη θα έχουν πια στα χέρια τους μόνο 60% της συνολικής ενέργειας για να αποφασίζουν. Και ερχόμαστε τότε λοιπόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο με συμμετοχή, με βούληση και γνώση των χωρών μελών. Ίσως αυτά να μην αρκούν σε, σε ορισμένους, αλλά χωρίς αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας που δεν θα ήταν ρεαλιστικό τώρα βλέπουμε ότι θα έχουμε 35% μετά θα έχουμε 40% δηλαδή μια σαφέστατη εξέλιξη των αρμοδιοτήτων προς την κατεύθυνση περισσότερου ευρωπαϊκού ελέγχου και περισσότερου ευρωπαϊκού επίπεδου. Εάν λοιπόν τώρα αυτό το σενάριο, εξετάσουμε αυτό το σενάριο των ανανεώσιμων ενεργειών, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στις χώρες μέλη. Ε, μεγάλη ε, χώρα, η Πολωνία, ας πάρουμε για παράδειγμα, όπου 90% του ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται 90% από άνθρακα. Δεν το θεωρώ πιθανόν και ρωτώ και τους παρόντες βουλευτές όλων των κομμάτων αυτής της μεγάλης αναπτυσσόμενης ε, οικονομικά χώρας της Πολωνίας. Θεωρείται ότι η πολιτική ανεξαρτήτως κυβερνήσεων θα θέλει να μειώσει στο 0% ή μετάσχει προς το 0% την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από άνθρακα. Δεν το πιστεύω. Και στην Πολωνία σχεδιάζεται νέος πυρηνικός σταθμός. Δηλαδή οι Πολωνοί εταίροι θέλουν να συμβάλλουν με πυρηνική ενέργεια στο energy mix τους έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο και επομένω από τη ρωσική κοινοπολιτεία. Μα, κυρία Χάρμς, αυτή η κυβέρνηση είναι δημοκρατικά εκλεγμένη. Και ειδικά εμείς οι Γερμανοί δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα καλύτερα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι οι Πολωνοί φίλοι έχουν υπόψη τους, έχουν συνείδηση για τις ανάγκες ασφάλειας, ασφάλειας το ίδιο όπως όλοι, και, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε λίγο την τάση, αγαπητέ κύριε Σούλτς, εμείς από τη, από τη Γερμανία να προσπαθούμε να θέλουμε να κατευθύνουμε ολόκληρη την κίνηση στην Ευρώπη και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο μετριόφρονες, πιο μετριοπαθείς και να δεχόμαστε και τις διαφορετικές του απόψει που υπάρχουν στην Πολωνία και στη Γαλλία. Το επόμενο, παρατηρήσει Σούλτς χωρί μικρόφωνο. Ομιλώ ω Ευρωπαίο απαντά ο κ. Σέτιγκερ, ο οποίο γνωρίζει την χώρα του, τη Γερμανία και που έχει μεγάλο σεβασμό για τι δημοκρατικέ διαδικασίε στην Πολωνία, Γαλλία και σε όλε τι άλλε χώρε μέρη. Και γι' αυτό ξαναλέω, όποιο έχει 90% παραγωγή ρεύματο από άνθρακα, δύσκολα θα καταφέρει να το κατεβάσει στο μηδέν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο σχεδιασμό, στον σχεδιασμό, ο άνθρακα, εάν δεν υπήρχε θέμα ε, διοξιδίου του άνθρακα θα ήταν διαφορετικά. Όποιο γνωρίζει την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, πρέπει να αφήσει χώρο και για τον άνθρακα στην ε, Ευρώπη του 2020. Η ΔΕΜΗ θα αντιμετωπίσει προβλήματα με ε, δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια και κυβερνήσεις. Γιατί υπάρχει και ο άλλος στόχος του διοξιδίου του άνθρακος που πρέπει να μειωθεί τις επόμενες δεκαετίες. Εδώ, σε συνεργασία με την Επίτροπο Χέντεγκαρτ, έχουμε προβλέψει 10% λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακο για τα επόμενα χρόνια σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. Σα παρακαλώ μην διακόπτε τον Επίτροπο. Όσον αφορά τώρα τα πυρηνικά εργοστάσια, συνεχίζει ο κύριος Έτιγκερ, γνωρίζετε και γνωρίζω ότι υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν τώρα μορατόριο για την ε, χρησιμοποίηση των πυρηνικών εργοστασίων ή που σκοπεύουν να τα κλείσουν άλλες γειτονικές χώρες όπως η Ελβετία. Αλλά υπάρχουν και άλλα που κτίζουν πυρηνικά εργοστάσια. Βλέπετε Φιλανδία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικά εργοστάσια και φτιάχνουν και άλλα και άλλες που δεν έχουν και πρόκειται να αρχίσουν να φτιάχνουν. Γι' αυτό και βρίσκω ότι είναι σημαντικό ανεξάρτητα από όλες αυτές τις διαφορές και τις διαφορές νοοτροπιών να γίνουν οι δοκιμασίες αντοχής με τα ύψιστα δυνατά επίπεδα ε, κριτηρίων ασφαλείας και να γίνει δεκτό αυτό από όλες τις χώρες μέλη. Πρόκειται για έναν μικρό, ελάχιστο βέβαια, αλλά κοινό παρονομαστή. Για χώρες λοιπόν που έχουν πυρηνικά εργοστάσια και χώρες που δεν έχουν. Και λέχθηκε ακόμη ότι η αρχή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Κυρίε και κύριοι, σε διάφορους τομείς της ζωής έχουμε δημόσιους ελέγχους για την υγεία, για την ασφάλεια, για τη τροχιά κυκλοφορία για την βιομηχανία, για την ενέργεια και ούτω καθεξής. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον δημόσιο έλεγχο. Και κυρία Χάρμς, όταν μιλάτε για κύκλους γνωστών, εάν όμως δεν είναι... Διακόπτη κυρία Χάρμς. Κυρία Χάρμς, βρίσκω ότι πρόκειται και για έκφραση δυσπιστίας από πλευρά σας απέναντι στον συνάδελφό σας κύριο Τριτίν, ο οποίος ήταν υπουργό Ενέργειας στην Γερμανία για 7 χρόνια. Εγώ έχω καταρχήν εμπιστοσύνη στις αρχές εποπτείας και καταρχήν πρόκειται να συνεργαστούμε μαζί τους και θα σας υποβάλω σε πλήρη διαφάνεια το σχέδιο για, την, ε, για τις δοκιμασίες αντοχής με την ελπίδα να λάβω από εσά προτάσεις διόρθωσης και βελτίωσης έτσι ώστε εν τέλει να υπάρξει ευρία αποδοχή από πλευρά όλων των χωρών μελών και πυκνότητα ελέγχων. Για πρώτη φορά με αυτές τις δοκιμασίες αντοχής που μας ζήτησαν να αναλάβουμε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, έχουμε στην πραγματικότητα μια κοινή ευρωπαϊκή διαδικασία για εξασφάλιση ύψης της ασφάλειας όλων των πυρηνικών εργαστασίων και αυτό αποτελεί μια καινοτομία και μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια τελευταία ερώτηση. Εγώ πήρα από τον Ιούνιο 2009 μια οδηγία η οποία πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τον Ιούλιο φέτος και σας λέω καθαρά δεν μου αρκεί σε ό,τι αφορά την ουσία της η οδηγία αυτή. Διότι πρόκειται κυρίως για τυπικές αριθμίσεις, καθορισμό αρμοδιοτήτων, υποδείξεις προς τις αρχές, αλλά επί της ουσίας δεν αρκεί. Και γι' αυτό παράλληλα με, τις, ε, με τους έλεγχους ασφαλείας και μέσα στα πλαίσια πάντοτε της εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητήσω μαζί σας και πώς μπορούμε σύντομα να αναθεωρήσουμε την οδηγία αυτή και να δώσουμε, να, να προσφέρουμε ουσιώδεις ρυθμίσεις για, για το ευρωπαϊκό επίπεδο και τους ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Now, dear, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, μπλε κάρτα, γαλάζια κάρτα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διατυπώσετε ερώτηση προς τον Επίτροπο ή το Συμβούλιο, μόνο μεταξύ συναδέλφων. Γι' αυτό παρακαλώ μην κάνετε τον κόπο να σηκώσετε την πλεκάρτα για τον Επίτροπο ή για το Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκιούρη. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική η συζήτηση. Σας ευχαριστώ, την άκουσα πολύ ενδιαφέρον. Η Προεδρία της Ουγγαρίας